Good morning everybody. Καλημέρα σας, καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι έχουμε αρκετά μέλη για να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι η τελευταία μέρα της Επιτροπής για αυτή τη θητεία. Τελευταία μας συνεδρία είναι σημαντική ημέρα Έχουμε πλήρη ατζέντα, πολλές ψηφοφορίες και θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι, ότι στην αρχή του μεσημεριανού διαλύματος θα πάρουμε μία φωτογραφία των μελών. Και μετά το τέλος της συνεδρίασής μας θα ήθελα να σας καλέσω για ένα ποτό από χαιρετιστήριο. Πηγαίνουμε κατευθείαν στο 6. Βλέπω ότι η ατμόσφαιρα εδώ μέσα σήμερα είναι απέσια. Είναι, κάνει πάρα πολύ ζέστη στην αίθουσα και ελπίζω να γίνει σύντομα κάποιος να κάνει κάτι γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε στο 6 Corrigendum. Δίνω αμέσως το λόγο στον εισηγητή και μετά θα ψηφίσουμε. Άρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το κοριτζέντουμ, το διορθωτικό, έχει να κάνει με δύο τεχνικές τροπολογίες που απαιτούνται από τους γλωσσονομαθείς για να αποσαφενιστεί το κείμενο σε δύο άρθρα και για να ευθυγραμμιστεί με όσες συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο. Το 11α ε, εισαγάγει την, καλή, την ίση μεταχείριση ώστε να μπορούν να περάσουν οι από τη δεύτερη φάση στην τρίτη και με τον ίδιο τρόπο αποσαφηνίζει ότι οι κανόνες για τις ποσότητες των ε, πιστοτικών πόντων εφαρμόζονται για όλους. Τώρα έχουμε στο 24 του, της αρχικής οδηγίας, όχι της εκθεσής μου. Εδώ Βάζουμε την τροπολογία για την ε, επιτροπολογία ε, για να βάλουμε αυτό το οποίο ζητήσαμε σαν Ευρωκοινοβούλιο. Δεν δίνεται ρητός στην αναθεώρηση ETS. Πρόκειται για την τυποποιημένη επιτροπολογία και η διαδικασία με εξέταση θα είναι αυτή βασική διαδικασία όπως προβλέπεται στο Omnibus. Λοιπόν αυτές είναι δύο τεχνικές τροπολογίες που μας προτείνονται από τους γλωσσομαθείς νομομαθείς. Ευχαριστώ. Thank uh, Σας ευχαριστώ και εγώ. Είστε σαφείς. Ψηφίζουμε. Σας παρακαλώ ετοιμάσετε την κάρτα ψηφοφορίας. Θα χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονικό σύστημα. Υπέρ. Παρακαλώ. Α, άνοιξα το σύστημα, τώρα τα άνοιξα, εντάξει, συγγνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. The very first vote, I will wait a little bit. Θα περιμένω λίγο. Everybody had voted. Όλοι ψήφισαν. Όχι ακόμη. Okay. <laughs> The vote is closed. Έληξε ψηφοφορία. Έληξε τα, αποτελέσματα. 40 υπέρ, 0 κατά. Δεν υπάρχουν αποχές. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Αμρέλ. Περνάμε στο επόμενο θέμα, το 6α, άλλο διορθωτικό. Και δίνω το λόγο στον εισηγητή Γκρότε. Δεν τον βλέπω εδώ όμως. Yeah, I think that there are here no information about problems, so maybe let me adopt. Λοιπόν, να συγκρίνουμε το κοριτζέντουμ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ. Everybody had voted. Ψήφισαν όλοι. Έληξε ψηφοφορία. 37 υπέρ, κανείς κατά, καμία αποχή. Εγκρίθηκε. Σημείο 7. Καθηγητής Αντώνιος Τρακατέλης. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Όχι ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω συζητήσεως. Thank you very much, Professor. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ψηφίσετε. Ξεκινούμε με την τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 της κυρίας Ρης και 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22. Υπέρ, κατά, ηλεκτρονικά. Για το 22 της κυρία Σάρμπο. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. The vote is closed. Έληξη ψηφοφορία. 23 εγκρίνεται. 23 κρούπα Περ, κατά αποχές απορρίπτεται. 24 τρακατέλης και υπόλοιποι κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται αλλά ας το ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά έληξη ψηφοφορία 23 εγκρίνεται. 24 εγκρίνεται. Ήτρε 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 και 26 όμοιες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 δάμου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απεσύρθη το επόμενο 28 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά Ψηφίζουμε. Έλξη ψηφοφορία. 23 υπέρ, 19 κατά. Γκρίνεται. Ήτρε 6 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά προτιμώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Έλλειψη ψηφοφορία. 25 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Το επόμενο καταπίπτει 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 3, 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αποσύρθη το επόμενο έχουμε δύο ταυτόσιμες 34 και 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 προφορική τροπολογία ρης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 310 καταπίπτει Παρα... 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται διαδικαστικό οι επόμενες τρεις τροπολογίες 38, 11 και 39 συνδέονται η δικιά μου τροπολογία γράφει ότι καταπίπτει αν το ΙΤΡΕ 11 εγκριθεί ε, το αμφισβητώ. Πιστεύω ότι είναι συμβατά και με το 38 και με το 11. Και θα ήθελα να το ψηφίσουμε ξεχωριστά, όπως προβλέπετε εδώ. Και σε λέξουν μετά οι υπηρεσίες και αν υπάρχει ένα πρόβλημα βλέπουμε. Πρόεδρος. Ωραία. Θα το ψηφίσουμε άσχετα από το 38 και μετά θα αποφασίσουμε τι θα κάνουν οι υπηρεσίες. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το επόμενο καταπίπτει 39 ντόιλ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία έλεξη ψηφοφορία 33 υπέρ 12 κατά εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ ακαταπίπτει 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 44. Έλξη ψηφοφορία. 33 υπέρ 13 κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει το επόμενο ήτρε 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 45 περ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Σημείο 1, τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε 1. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ήτρε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σχέδιο έκθεσης όπως τροποποιήθηκε τώρα ηλεκτρονικά ψηφίζουμε άρχεται ψηφοφορία έληξη ψηφοφορία 43 υπέρ 6 κατά δεν υπάρχουν αποχές το σχέδιο ψηφίσματος ηλεκτρονικά. Έληξη ψηφοφορία, 42 υπέρ, 7 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια καθηγητά κύριε Τρακατέλη. So let me move to item I. Προχωρούμε λοιπόν στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Βλέπω τον εισηγητή στην αίθουσα. Θέλετε το λόγο, θέλετε να κάνετε μια σύντομη δήλωση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι πριν από λίγες εβδομάδες συζητήσαμε τις τροπολογίες τις οποίες υπέβαλα σε αυτό το σχέδιο κανονισμού. Εν τω μεταξύ διεξήχθη ένα τρίλογος και με το Συμβούλιο. Είχαμε τρεις επίσημους ε, διαλόγους με το Συμβούλιο. Ε, δεν ήταν εύκολες αυτές οι διαπραγματεύσεις. Καταρθώσαμε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία κατόπιν στα πλαίσια της Κορεπέρα ακολούθησε μια συζήτηση. Ε, ξέρετε ότι η Τσεχική Προεδρία δεν υποστήριξε τις απόψεις του Κορεπέρ ε, και οι σκιώδεις εισηγητές ε, έκαναν μέτωπο θα έλεγα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πακέτο 40 τροπολογιών. Πρόκειται για συμβιβαστικές τροπολογίες και υπάρχει μια τροπολογία του κυρίου Χέγγι ήταν τελικά μια πολιτική συμβιβαστική τροπολογία στην οποία καταλήξαμε και έτσι μπορέσαμε να διασώσουμε τα σημαντικότερα στοιχεία της πρώτης ανάγνωσης και προσπαθούμε να υπάρχει συνέπεια ε, να συνάδουν τελικά οι στατιστικές σχετικά με τα ζυζανιοκτώνα ε, και με τους άλλους κανονισμούς που αναφέρονται στην αηφόρο ανάπτυξη και στην ε, εμπορία αυτών των προϊόντων. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη ένα νέο κανονισμό που αναφέρεται στον τρόπο της χρήσης των στατιστικών. Υπάρχει μια συμφωνία ε, με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή. Αν υπάρξουν νέες συμφωνίες για τα βιοκτώνα θα δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Θέλουμε να υπάρξει μια μελέτη για τις συνέπειες της εφαρμογής αυτής, της, αυτού του κανονισμού και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί τελικά μπορώ να υποστηρίξω αυτή την συμβιβαστική τροπολογία την οποία υποστηρίζουν όλες οι πολιτικές ομάδες Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε κάνει πολλά βήματα προς τα μπρος σε σχέση με την νομοθεσία και μετά από την έγκριση στην Ολομέλεια μπορούμε να έχουμε ε, τελικά μια νομοθεσία τον Απρίλιο, το αργότερο τον Μάιο. Ο Πρόεδρος, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι δεν είναι υποχρεωμένοι οι σκιώδες εισηγητές να κάνουν δηλώσεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Όπως γνωρίζετε, θα ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία η οποία περιλαμβάνει τις 40 πρώτες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, καταπίπτουν οι επόμενες δύο, και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την, ε, το σχέδιο συστάσεων. Άρχεται η ψηφοφορία. Περιμένουμε την Άνια Πασκιόρμπε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίας. 47 υπέρ, μία αποχή και ένας κατά. Ε, ένας κατά και καμία αποχή. Πολύ ωραία, χαίρομαι. Συγχαρητήρια. Προχωρούμε τώρα και θα ασχοληθούμε με τον πιο δύσκολο φάκελο στην ημερήσια μας διάταξη σήμερα. Μιλούμε για την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Να δώσω το λόγο στον Τζον Μπόις για μια σύντομη δήλωση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντω θα είναι σύντομη η δήλωσή μου, διότι μπορείτε να έχετε τη μεγάλη εκδοχή των πραγμάτων και τη σύντομη, την βραχή εκδοχή των πραγμάτων. Διανύσαμε μεγάλη απόσταση ως προς το θέμα αυτό. Ως Επιτροπή στην αρχή ασχοληθήκαμε με την έκθεσή μας για την κινητικότητα των ασθενών και όλα αυτά έγιναν πριν από τρία χρόνια, αν όχι και περισσότερα. Και καταφέραμε η έκθεση αυτή να υποβληθεί στην Ολομέλεια. Τώρα έχουμε ασχοληθεί με τις συνέπειες των νομικών διαδικασιών που ακολουθούνται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θέλουμε δηλαδή να προσφέρουμε νομική ασφάλεια και διαδικαστική σαφήνεια στις προτάσεις αυτές. Ελπίζω ότι καταφέραμε να βελτιώσουμε το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να πω ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία ήμασταν σε στενή επαφή και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο με την αντίστοιχη Προεδρία του Συμβουλίου, πρώτα με τη Γαλλική Προεδρία και τώρα με την Τσεχική. Και είμαι ευγνώμων στους, για τους ε, επιτετραμένους για θέματα υγείας των ε, δύο Προεδριών του Συμβουλίου, οι οποίοι πολύ συχνά με επισκέφτηκαν. Ο σκοπός μας ήταν να καταλήξουμε σε μια πρόταση η οποία να καλύπτει τις ανάγκες τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των κρατών μελών. Από εκεί και πέρα, όποια έκβαση και αν έχει η ψηφοφορία, εγώ θα ήθελα πάντως να ευχαριστήσω θερμά από τα βάθη της καρδιάς μου τους συναδέλφους μας στην Επιτροπή. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικώς κύριε Πρόεδρε για τη δουλειά σας και θέλω να ευχαριστήσω πάνω από όλους τους σκιώδεις εισηγητές διότι πραγματικά κόπιασαν για να πετύχουμε τους στόχους μας. Κόπιασαν διότι έπρεπε να λάβουν υπόψη τους τις ανάγκες των δικών τους συναδέλφων από τις άλλες ομάδες, παραμένοντας όμως ανοιχτοί στις απόψεις των υπολείπων. Ευχαριστώ τους δικούς μου συναδέλφους, αλλά και όσους είναι εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τροφοδότησαν αυτή τη συζήτηση με χρήσιμες ιδέες. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό μου, τους βοηθούς μου, τον Νίλ και τον Μάρκ, οι οποίοι δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά, μαζί με το προσωπικό τους βοηθούς των ε, σκιωδών εισηγητών και των συντακτών γνωμοδότησης από άλλες επιτροπές. Ξέρετε, πολύ συχνά ε, φορτώνουμε τους ώμους των βοηθών μας με εξαιρετικά μεγάλο βάρος και έχει έρθει η στιγμή να τους χειροκροτήσουμε και να τους ευχαριστήσουμε θερμά για την πολύ σκληρή δουλειά τους. σίγουρα το αξίζουν, αξίζουν τα συγχαρητήριά μας. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συμβούλους που είχαμε, την Ζαγαλντίν, στη δική μου περίπτωση, η οποία μας βοήθησε πολύ. Αλλά επεκτείνω τις ευχαριστίες αυτές σε όλους τους συμβούλους που μας έχουν βοηθήσει είτε παρασκηνιακά είτε στο προσκήνιο. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω θερμά και μία κυρία η οποία υποτίθεται ότι δεν είναι πια μαζί μας, αλλά παρόλα αυτά μέσω ε, γραμματείας ε, έχει αναλάβει τα καθήκοντά της και τα συνεχίζει να τα διεκπεραιώνει παρόλο που δεν είναι στη γραμματεία. Την βλέπετε πάνω στο πάνελ, την Βεατρής. Ε, έχει έρθει η ώρα λοιπόν να ψηφίσουμε. Ευχαριστώ. Πήρετε τα λόγια από το στόμα μου και εγώ αυτό ακριβώς ήθελα να τονίσω. Ήθελα να πω ότι όντως φεύγει η γιατρής. Δεν θα είναι πια μέλος του διοικητικού προσωπικού της Επιτροπής μας. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να την ευχαριστήσουμε θερμά εξ ονόματος των μελών όλες της Επιτροπής για τη δουλειά της. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία θέλω να πω και εγώ δύο λόγια, διότι ξέρετε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η διαδικασία, πόσο πολύ παλέψαμε για να αναγνωριστούν οι αρμοδιότητες μας για το θέμα αυτό βάσει του κανόνα 47 για την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Και γι' αυτό επί τη βάση του κανόνα 47 αποφάσισα να ενσωματώσουμε τις τροπολογίες 55, 56, 64, 65 και 66 από πλευράς Επιτροπής για την απασχόληση και τις τροπολογίες 8, 9, 10 και 11 από πλευράς Επιτροπής για την εσωτερική αγορά. Κάποιες από τις δεύτερες, οι 8, 9 και οι 10, δεν είναι συμβατές με την 110 και την 113, οι οποίες στοχεύουν στη διαγραφή των αιτιολογικών σκέψεων τα, οι υπόλοιπε μπορούν να, προσθεθούν ως, να ψηφιστούν ως προσθήκες χωρίς ε, περαιτέρω ε, τροποποιήσεις. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Ήταν πολύ περίπλοκη αυτή η διαδικασία. Επιμένω ότι εγώ πήρα προσωπική απόφαση για τροπολογίες που δεν σχετίζονται με το εγγενές πνεύμα, αν θέλετε, το περιεχόμενο της έκθεσης. Ξεκινούμε λοιπόν με την τροπολογία υπαριθμών 42, 43 και 44 οι οποίες στοχεύουν στην απόρριψη της πρότασης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Σαρανταεννέα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 και 47-1 από την Επιτροπή Γυναικών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 51 και 52 μαζί υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρα της ψηφοφορίας. 22 υπέρ, μία κατά απορρίπτε. Ε, εγκρίνεται. 46. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική υπαριθμόν 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Ενοποιημένη τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά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 Ας κάνουμε ένα άλμα. Πάμε στη σελίδα 7, αν δεν απατώμε. Να ψηφίσουμε την τροπολογία του κυρίου Μπλόκλαντ και της κυρίας Ντάλ. Την τροπολογία 2.15. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο ίδιες. Οι 2.17 και οι 2.18. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές, ας ψηφίσουμε ε, με το ηλεκτρονικό σύστημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 29 κατά, απορρίφθηκε. Απορρίπτονται. 2.19. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.20, 2.21, 2.24 και τις τρεις μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Οι 2.22, οι 29 της Επιτροπής Απασχόλησης και οι 6 της Επιτροπής Οικονομικών είναι ίδιες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, για να το επαληθεύσουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραστη της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 20, 27 κατά. Απορρίπτονται. 2, 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2, 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε παρακαλώ. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Πενήντα υπέρ. Κανείς κατά. Μάλλον παραπλανήθηκα λόγω του του σερβιρίμισματος του τσαγιού και νομίζω ότι ήταν περισσότεροι κατά. 2.26. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο ίδιες. Οι 2.27 και οι 2.28. Αλλά και οι 30 είναι ίδια. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Οι επόμενες δύο καταπίπτουν Ας πάμε στην 7 έκον. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας πάμε στην επόμενη σελίδα. Θα ψηφίσουμε αυτή είναι αργότερα. Πάμε στην 2.38 και τη 2.39. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Η επόμενη καταπίπτη 2.41 του κυρίου Ζίμπερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.42 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η επόμενη καταπίπτη. Ήμκο 24 στη δική μου σελίδα 11. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 33 κατά. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώς παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 25 υπέρ. 32 κατά. Απορρίπτεται. Έχουμε κάποιες που είναι ίδιες. Η 255, η 256, η 257, η 258, η 11 του Ήτρε, 13 του ΦΑΜ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Οι επόμενες δύο καταπίπτουν. 2.61 και 2.62 είναι ίδιες. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές εγκρίνονται. Η επόμενη καταπίπτη 263 των Τούρμες και Άουκεν. Και αυτή καταπίπτη 264 Σορνόθα Μαρτίνεθ και Αγιάλα Σέντερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 265 σύνοτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρεις ίδιες, οι 266, οι 267 και 25 ίμκο, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 268. Εστρέλα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 269. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 270. Εστρέλα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 271, 272, 2.73, 274 και 275. Όχι. Μέχρι και τη 275. Τις ψηφίζουμε μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Η επόμενη καταπίπτει. 277. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δύο ίδιες οι 2.78 και οι 12 ήτρε. Ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τρεις ίδιες. 2.79, 12 έκον και 36 employment. Ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνονται. 2.81 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 280, ΙΜΚΟ 26, υπέρ. Κατά. Αποχές να το επαληθεύσουμε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. «24 υπέρ, 30 κατά, απορρίπτεται». «282, ποιος είναι υπέρ» κατά, αποχές, απορρίπτεται. 283 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, υπέρ. Το 37 κατά, αποχές, εγκρίνεται, δύο ίδιες. Οι 284 και 27 ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 286 ίδια με 29 ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Πάλι δύο ίδιες, 2,85 και 28 ΙΜΚΟ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 2,87 και 2,88. Ήταν οι ίδιες με τις προηγούμενες που ψηφίσαμε. Επομένως έχουν εγκριθεί ήδη. Πάμε στην 2,89 και στην 2,90. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 2,92 και 38 employment. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτονται. 2.92 υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. John Bowies, 2.92. Πέρας της ψηφοφορίας. 44 υπέρ, 7 κατά μία αποχή. Εγκρίνεται. 2.93. Καταπίπτει. Πάμε στην 300. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 301 και 377. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 3.02 και 13 ήτρε υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραστη ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 35 κατά. Απορρίπτονται. Να ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 305, η οποία εν μέρη καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία 5, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε το υπόλοιπο. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 5. Τροπολογία 303 μαζί με τη 14 Ήτρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Κάποια ευτυχή ε, δευτερόλεπτα διαλύματος για μένα. Μέχρι να βρω τη σελίδα 25 στο δικό μου κατάλογο ψηφοφοριών. Έχουμε χρόνο. Μπορούμε να προχωρήσουμε πιο αργά. Τρία 61 είναι η τροπολογία που θα ψηφίσουμε τώρα. Ίδια με την 35.2 της ΣΥΜΚΟ. ψηφίζεται ως αιτιολογική σκέψη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 της στην ίδια σελίδα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Κατά 35-7 της ΙΜΚΟ. Υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 30 υπέρ 26 κατά. Εγκρίνεται. Έκον 13 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 366 υπέρ, κατά, αποχές. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώς παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 366. Πέρας της ψηφοφορίας είναι σαφής η απάντηση. 48 υπέρ, 7 κατά. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Η 367, 368, 369, 370 και οι 18 της Ήτρε είναι ίδιες. Τις ψηφίζουμε μαζί όλες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 371. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώς παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. 371. Ψηφίζουμε την 371. Πέρα της ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 31 κατά. Απορρίπτεται. Ήμκο 36. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Να τα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώς παρακαλώ. ΙΜΚΟ 36. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας, 26 υπέρ, 28 κατά μία αποχή. Απορρίφθηκε. Προς Προσψήφιση. Ίδια με 373. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. «3.74. Αντρέγευς. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3.76. 49 της employment, 15 έκον, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 378 υπέρ. Κατά, αποχές, να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικώς παρακαλώ. Την 378 ψηφίζουμε. Πέρα της ψηφοφορίας 26 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. 379 Μακέιβαν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει. Η επόμενη καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία. Πάμε στη σελίδα, στη σελίδα 29. Έχουμε την 20 της Ήτρε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη σελίδα 33. 4.17 για την καινούργια παράγραφο 3α του άρθρου 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Πάμε στη σελίδα 35. Ψηφίζουμε την 425 της κυρίας Μπρόπελς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 426. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι επόμενες δύο θα ενσωματωθούν αμέσως. Ήτρε 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4.27, 4.28 και 4 και 23 της Ήτρε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 4.30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4.32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.34 και 4.35 για τη διαγραφή του άρθρου 7 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.38 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Δύο ίδιες. Η 436 και η 42 ΙΜΚΟ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 57 της employment. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρθρο 7. Παράγραφος 1α καινούριο. Τροπολογία της κυρίας Σίνω. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4.40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι επόμενες καταπίπτουν. Γι' αυτό πάμε στην 4.42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δύο ίδιες. 18 και 43 ήμικο υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Προχωρούμε τώρα. Και πάμε στη σελίδα 40. 467 τροπολογία. Ε, εσείς το έχετε στη σελίδα 39 νομίζω. 467. 467 τροπολογία. Στην, ε, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα μπορούσαμε τώρα να πάμε στη σελίδα 42. Μιλώ για την 481 των Τούρμες και Άουκεν για το παράγραφο 4 του άρθρου 8. 3α μάλλον του Άρθρο 8. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στην επόμενη σελίδα. Στη σελίδα 43. Έχουμε μία τροπολογία η οποία έχει ενσωματωθεί αμέσως και δεν ψηφίζουμε την 21 ΦΕΜ. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 44, στην τροπολογία 4-4-3-5 σε παρέθεση. Τροπολογία της κυρίας Φερέιρα και λοιπόν, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Είναι στη σελίδα 43 στο δικό μας κατάλογο ψηφοφοριών. Τροπολογία 443. Σε παρένθεση 5. Πέρα της ψηφοφορίας. 23 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. Προχωρούμε τώρα και πάμε στην 494 του κυρίου Φιέλνερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για να δούμε τι θα κάνουμε με την επόμενη τροπολογία. Καταπίπτει ή όχι. Καταπίπτει. Καλώς. Πάμε σε δύο ίδιες. Την 495 και 29 ήτρε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 22 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει. Πάμε στο άρθρο 8, παράγραφος 5α, β και γ. Καινούρια διατύπωση. 497 της Τζούλα Χέτζη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 498. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι επόμενε δύο είναι ίδιε. 4,99 και 31 ήτρε. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να το δούμε ηλεκτρονικώ. Ψηφίζουμε δύο ίδιε τροπολογίε, Την 4,99 και την 31 τη ήτρε. Πέρα τη ψηφοφορία, 32 υπέρ. 23 κατά. Εγκρίνεται. Οι επόμενες καταπίπτουν. 5.01. Υπέρ κατά. Αποχές απορρίφθηκε η 501. Ήταν ε, ταυτόσιμες. Ήμκο 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Έχουμε δύο ταυτόσιμες. Την 22 και την 503 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η επόμενη που πρέπει να ψηφιστεί 67 υπέρ κατά αποχές Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης, η 67 ψηφίζεται, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Λοιπόν, 56 υπέρ, 23, 23 ε, υπέρ, 32 κατά, απορρίφθηκε. 504 και 249 υπέρ, κατά, αποχές ας το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά 504 και ΙΜΚΟ 49 άρχεται πέρας της ψηφοφορίας 33 ήταν υπέρ 20 κατά εγκρίθηκε ...505 και ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε έχουμε δύο ταυτόσημες όχι όχι μόνον, την έκον 21 έχουμε υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 464 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 509 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 5-6 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 5-0-9 και η 43 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε και τώρα έχουμε τρεις ταυτόσιμες Πέντε δώδεκα. Συγγνώμη, συγγνώμη. 5.08 πρέπει να ψηφίσουμε αυτήν τώρα. Είναι σαφές, έκανα ένα λάθος. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίφθηκε. Τώρα έχουμε τις τρεις ταυτόσημες, 512, 68 και 22. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκαν. 513 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τώρα, στην επόμενη σελίδα έχουμε το άρθρο 9, παράγραφος 2, καινούρια. Νέα, έχουμε την 517 Βέστλοντ υπέρ κατά αποχές, απορρίφθηκε 517. 518 και 519 είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκαν. Τώρα, οι επόμενες δύο εκπίπτουν. Το ίδιο και οι επόμενοι. 522 no vote. Δεν την ψηφίζουμε. Η επόμενη είναι η 525. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε ο 825. Λοιπόν, στην περίπτωσή μου θα αλλάξω σελίδα και θα έχουμε τη σελίδα 47, έχουμε 538, λοιπόν είναι σαφές ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές απορρίφθηκε 538 βουτιερές Κορτινές 539 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 541 υπέρ «539 θα την ψηφίσουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 45 ήταν υπέρ και 7 κατά. Λυπάμαι, αρχίσατε να κουράζεστε. Είναι διαφορετική κατάσταση από ό,τι προηγουμένως. Λοιπόν, εγκρίθηκε 539 και μάλιστα σαφώς. 541 υπέρ. Κατά. Ας το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας 24 υπέρ 27 κατά. Απορρίφθηκε. Τώρα έχουμε δύο ταυτόσημες. Την 540 και την 508. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκαν. 542 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Λοιπόν, έχουμε τις ταυτόσημε 24 και 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν. 543 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 544 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Στη σελίδα 50 Έχουμε την ΙΜΚΟ 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Στην ίδια σελίδα, εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης, 75 υπέρ, κατά, αποχές. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Έχω την εντύπωση ότι εγκρίθηκε 75, αλλά στο επαληθεύσουμε. Λοιπόν, 75 της Επιτροπής Απασχόλησης στο άρθρο 10, παράγραφος 2, α νέα. Νέο. Λοιπόν, πέρα της ψηφοφορίας ψηφίσατε όλοι. 32 ήταν υπέρ και 19 κατά καμία αποχή. Επομένως εγκρίθηκε. 252 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 555 εκπίπτει. 556 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Η επόμενη υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 557 έχει εκπέσει. Ήτανε ταυτόσημα μη με την 35. Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα τώρα. Όχι, όχι. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Γιούρι 5. Υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 58. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Γιούρι, της, 6. Υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Ε, απορρίφθηκε 22 υπέρ, 30 κατά η, της Γιούρι 7 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Στο άρθρο 12 τώρα έχουμε την 559 της κυρίας Κρούπα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 562 υπέρ κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία 562. Τροπολογία της κυρίας Φερέιρα, 562. Πέρας της ψηφοφορίας, 25-34 κατά απορρίφθηκε, 560. Κόρμπεϊ, υπέρ, κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, Ίσως να είναι η ίδια κατάσταση με την προηγούμενη, αλλά πρέπει να το επαληθεύσουμε. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Επαληθεύουμε την 560. Πέρας της ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 33 κατά, απορρίφθηκε. 561, 77 και 24 είναι ταυτόσιμες. Υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίθηκαν. 563 και ΙΜΚΟ 56 είναι ταυτόσιμες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκαν. Απασχόληση 78, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. ΙΜΚΟ 57, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τώρα μπορούμε να περάσουμε ορισμένες σελίδες. Στην περίπτωσή μου γυρίζω στη σελίδα 55 έχουμε το άρθρο 12 παράγραφος 2 πρόκειται για μια καινούρια παράγραφο α πέντε θα ψηφίσουμε πρώτα υπέρ κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Πέντε νέα τέσσερα υπέρ κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 596 Ούλμερ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 597 υπέρ κατά αποχές Απορρίφθηκε. Λοιπόν, στην περίπτωσή μου περνάω στη σελίδα 60, 15 1. Λοιπόν, 5 5-4-6 Ούλμπερ, υπέρ, κατά. Αποχέσα απορρίφθηκε 6.47 και επιτροπή Απασχόληση 96 υπέρ κατά θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας η 29 ήταν υπέρ και 24 κατά εγκρίθηκε 648 Φερέιρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 649 Λίζε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 650 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 651 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 652 υπέρ, κατά, εποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά ας το επαληθεύσουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε τις ψηφοφορίας, 27 ήταν υπέρ και 25 κατά, εγκρίθηκε. 653 υπέρ κατά αποχές ας το επαληθεύσουμε ψηφίσουμε την 653 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας 23 ήταν υπέρ 23, 33 κατά απορρίφθηκε Τώρα έχουμε τρεις ταυτόσημες, την 654 της 38 και 655. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκαν. Απασχόληση 99. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το επαληθεύσουμε. Της Επιτροπής Απασχόλησης Τροπολογία Υπερθμών 99. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 23 ήταν υπέρ, 32 κατά, απορρίφθηκε. 100 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ, κατά, αποχές. Ναι, ήταν η πλειοψηφία. 656. Weisgerber Ulmer, υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίφθηκε. 660 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 661 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 659 εκπίπτει, εκπίπτει, ναι, εκπίπτει 657 επίσης Η 661 την ψηφίσαμε την 661. Ψηφίσαμε την 661 αλλά εάν θέλετε μπορούμε να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Αντρέγευς. άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 30 ήταν υπέρ, 24 κατά. Εγκρίθηκε. Οι επόμενες δύο εκπίπτουν. Λοιπόν, ψηφίζουμε την Ρίπορς Ripples, υπέρ, κατά, Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας, 25-34 κατά μία αποχή, σαφέστατα απορρίφθηκε. Και τώρα οι επόμενες τρεις είναι ταυτόσιμες 663, 657 και 658 και ΙΜΚΟ 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκαν. Η επόμενη εκπίπτει. Τρεις ταυτόσημες. 34, 664 και ήτρε 39. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκαν. 665 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 666 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 667 υπέρ. Κατά. Ας το επαληθεύσουμε. 667. 667. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 31 κατά, απορρίφθηκε. 668 και 70 τη ΣΥΜΚΟ, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίφθηκε. 669 τούρμες όκεν, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίφθηκε. 670 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 670 671 671 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Δύο ταυτόσημες 672-673 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε, απορρίφθηκαν. 674 και 97 της Επιτρο... υπάρχει διαδικαστικό η κυρία Ρόμαν Βίτεν. Πρόεδρε, έχω μια προφορική τροπολογία. μπορεί να διορίσει η Επιτροπή ε, τους ειδικού ώστε να γίνεται ανάλυση, αξιολόγηση κλπ. Το έχετε και σε γραπτή μορφή, λέει ο Πρόεδρος. Είναι η προφορική τροπολογία στο άρθρο 15α, το καινούριο και στην τροπολογία 674 και 97 employment και έκον 28 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 675 και ήτρα 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Απορρίπτεται, απορρίπτεται, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Φέλνα σήκωσε μόνο το χέρι του. Εγώ έκανα λάθος, γλωσσικό λάθος. Λυπάμαι. 6-7-6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. 24 υπέρ 29 κατά απορρίφθηκε. Έσπασε, τι έσπασε. Κάτι ψιθυρίζει ο πρόεδρος, αλλά δεν ακούσαμε το σύνολο της φράσης. Τροπολογία 35 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επόμενη καταπίπτη και πάρα επόμενη καταπίπτη. πάμε στην 6, 7, 9 υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά 679 Έληξη ψηφοφορία. 22 υπέρ, 31 κατά, απορρίπτεται. 680 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές, κρίνεται. Employment, καταπίπτει. Πάμε στο ΙΜΚΟ 71 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται καταπίπτει και η επόμενη πηδάμε δύο σελίδες στο πάμε στη σελίδα 64 άρθρο 18 παράγραφος 1 employment 102 υπέρ κατά αποχές Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. 23 υπέρ, 29 κατά απορρίπτεται. Ήμκο 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Employment 103 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 698. Βάις Πέρβερ και Ουλμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ήμκο 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δύο όμοιες 699 και employment 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 700 Φερέιρα υπέρ κατά αποχές Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, έληξε 25 υπέρ, 31 κατά, απορρίπτεται. 701 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 702 υπέρ, κατά, αποχές, Λοιπόν, ηλεκτρονικά, δεν βλέπω πολλά χέρια. 702 λοιπόν. Έλξη ψηφοφορία. 34 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. Ήμκο 80 με προφορική τροπολογία εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ημκο 81 υπέρ κατά στο ελέγξουμε και ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία έληξη ψηφοφορία 16 υπέρ 39 κατά απορρίπτεται σαφέστατα 703 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 704 και employment 105 και έκον 29 όμοιες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 705 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 706 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται πάμε στην αιτιολογική έκθεση 53 υπέρ διαδικαστικό παρακαλώ Είχα στείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, αλλά ίσω καλύτερα να το διευκρινίσω εδώ. Υπάρχουν κάποιε τροπολογίες για τα σημεία του σκεπτικού της αιτιολογικής έκθεσης ε, ε, ε, και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι δεν υπάρχει αντίφαση. Η τροπολογία 60 αποσύρεται και η τροπολογία 87 ε, για αυτήν αποσύρεται το δεύτερο τμήμα που λέει δεν προδιαγράφει για τα κράτη-μέλη κτλ. Είχα στείλει αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικό, ηλεκτρονικά, αποσύρουμε λοιπόν το 60 και το δεύτερο μέρος του 87, της 87 μάλλον. Yeah, okay, Ωραία. Ελπίζω να κατάλαβα σωστά από τη διερμηνία. Ναι, τα στείλατε γραπτά, σωστό. Ε, θα του πηδήξουμε λοιπόν στο συγκατάλογο της ψηφοφορίας, εντάξει. Συμφωνείτε. Λοιπόν, περνάμε στην ετρολογική έκθεση. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η επόμενη καταπίπτη 57. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έκον 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Ψήφισαν όλοι. Έλεξη ψηφοφορία. 21 υπέρ 32 κατά απορρίπτεται. Η επόμενη αποσύρθηκε, όπως μας το είπε ο κύριος Λίζε, ΙΜΚΟ 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Employment 1 υπέρ κατά αποχές για να το ελέγξουμε πάλι ηλεκτρονικά. Chris Davis ψήφισε και υπέρ και κατά και μπερδεύτηκα γι' αυτό. Έλξη ψηφοφορία. 20 υπέρ, 35 κατά. Είναι σαφές το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Employment 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Employment 3, 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 για το σημείο 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η επόμενη καταπίπτει έκον 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται employment 4-5 4 και 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται employment 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά στο λέξουμε και ηλεκτρονικά αυτό The vote is closed. ψηφοφορία 25 υπέρ 30 κατά Employment 7 ίδια υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Employment 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Employment 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 τίσεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 Δύο ψηφοφορίες γι' αυτό. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου μέρους. Υπέρ του πρώτου μέρους. Κατά. Ας το ελέξουμε ηλεκτρονικά. Πρώτο μέρος της τροπολογίας 65, ΙΜΚΟ 2, είναι ταυτόσιμες. Έλεξη ψηφοφορία. 34 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος της 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ελέγξω το δεύτερο μέρος της ψηφοφορίας για το, την 65 πάντα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. 24 υπέρ, 31 κατά. Απορρίπτεται. ΦΕΜ 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. ΙΜΚΟ 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. 16 υπέρ 40 κατά. Σαφέστατη απόρριψη. 66 κυρία Λεωτάρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ραπορτέρ 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει. Employment check. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 68 κυρία Λεωτάρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται employment 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 και 70 ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2,71 71 και 24 4 υπέρ κατά 71 και 24 4 καταπίπτει έτσι λέει, καταπίπτει αν εγκριθεί το 69. Σωστό, ότι εγκρίθηκε το 69, καταπίπτει. Το επόμενο είναι γλωσσική τροπολογία. Ας περάσουμε στο, λέει ο πρόεδρος και διακόπτη, για να ελέγξω κάτι, για να ελέγξω κάτι. Πού να πάμε. Το ΙΤΡΑ 2, στο ΙΤΡΑ 2, που αφορά το σημείο σκεπτικού 9. Όχι. Εντάξει. Οκ. Okay. Σελίδα 68 λέει ο πρόεδρος. Οι προηγούμενες καταπίπτουν. Λοιπόν, ήτρε 2 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Έληξη ψηφοφορία. 34 34-19 εγκρίνεται. 76 έξι της κυρίας Τάισον υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Employment 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 με προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 78 και φαμ 4, 4 μάλλον, καταπίπτει και η επόμενη καταπίπτει και η επόμενη και η επόμενη και πάμε στην 84 η 84 είναι η Εντάξει. Σύνοτ. Που είναι όμοια με την 85 της κυρίας Λιωτάρδη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχουμε τρεις όμοιες 86, 6 και 87. Η δεύτερη είναι του Πίτερ Λίζα για το δεύτερο μέρος, του 87, το οποίο έχει αφαιρεθεί. Ψηφίζουμε λοιπόν αυτές τις τρεις. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Το ελέγχουμε ηλεκτρονικά καλύτερα.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 η επόμενη καταπίπτει 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Φαμ 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται φαμ 6 υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά φαμ 6 άρχεται η ψηφοφορία έλεξη ψηφοφορία 21 υπέρ 34 κατά απορρίπτεται φαμ 7 υπέρ κατά Δεν βλέπω χέρια. Υπέρ. Φαμ 7. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το ελέξουμε. Employment 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Employment 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επόμενη καταπίπτει 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκόν 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται γιούρι 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται employment 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105, 106, 107, 108 ίδια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το επόμενο καταπίπτει 109. Κυρία Λιωτάρδη, πέρα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η επόμενη καταπίπτει. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται employment 16 υπέρ κατά απο, αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ employment 16 28 υπέρ, 26 κατά, εγκρίνεται. Με μικρή διαφορά. Λοιπόν, στην επόμενη. 112 και ΙΜΚΟ 113 μάλλον. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114. Αν θα ελέγξουμε το 113 ηλεκτρονικά καλύτερα. Το 113 ηλεκτρονικά. Της κυρίας Μακέιβεν. Έλεξη ψηφοφορία 23 υπέρ, 30 κατά, απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τρεις όμοιες 116, 17, 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 122 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 καταπίπτει 4 καταπίπτει 120 έχει ενσωματωθεί και η 125 πρέπει να θεωρηθεί, αν εγκριθεί πρέπει να θεωρηθεί σαν πρόσθετο σημείο στην εκλογική έκθεση. 125 λοιπόν, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 124 ή 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δύο όμοιες, 127 και employment 17 υπέρ, κατά, Α, όχι καταπίπτει, καταπίπτει, δικό μου λάθος λέει ο Πρόεδρος. Πάμε στο 128 και 129. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 130 υπέρ. 128 και 129 θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Έχουμε δύο όμοιες τροπολογίες, αριθμών 128 και 129. Τις ελέγχουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εντάξει, πρόκειται για την αιτιολογική σκέψη 26. Ψηφίσατε όλοι, έλξη ψηφοφορία. 25 υπέρ, 30 κατά, είχα δίκιο. 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 131 και 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήτρα 4 είναι το επόμενο. Έχουν ενσωματωθεί την προηγούμενη. Ήτρα 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το επόμενο έχει ενσωματωθεί με τον κανόνα 47. Πάμε στην 134 υπέρ. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται φέμ 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η επόμενη καταπίπτει και να ελέγξουμε την 138 καταπίπτει και αυτή Ήμκο 12. Υπέρ. Ήμκο 12. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Φεμ 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 139. Για να δω, για να δω. Ένα λεπτό, να συνεννοηθώ. Καταπίπτει. 141 Βάις Κέρμπερ ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δύο όμοιες 142 και 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται employment 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ καταπίπτει, καταπίπτει συγγνώμη λέει ο πρόεδρος και η επόμενη καταπίπτει έχουμε δύο όμες 145 και 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται employment 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, α, απορρίπτεται με συγχωρείτε 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Το 157 πάμε κατευθείαν. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Employment 20, υπέρ, κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Employment 20. Άρχεται η ψηφοφορία, έληξε κιόλας. 32 υπέρ 24 κατά εγκρίθηκε 158 υπέρ καταπίπτει mm. λάθος το φακελό μου 158 κατα... καταπίπτει γιατί εγκρίναμε το employment 20 και όχι 29 όπως γράφει το έγγραφό μου. 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 159. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 160. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Employment 21. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Employment 22. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 161 υπέρ Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Καταπίπτει 161. 156 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Εδώ για να το δούμε. 156 ψηφίζουμε. Έληξη ψηφοφορία 32 υπέρ 24 κατά. νεκρήθηκε. Το επόμενο καταπίπτει 162 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 164 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται η επόμενη καταπίπτει και πάμε στη 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε ΙΜΚΟ 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 172 σημείο 39 α νέο Πανεπιστημίου της αιτιολογικής έκθεσης παράγραφος. Υπέρ 172. Νέο σημείο στην αιτιολογική έκθεση 29. Υπέρ κατά απορρίπτεται. «173 και ΙΜΚΟ 17 ταυτόσιμες υπέρ» κατά για να το ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά λοιπόν ψηφίζουμε και έρχεται η ψηφοφορία. Έληξη ψηφοφορία. 27 υπέρ 30 κατά απορρίπτεται. 174 Weisberger Ulmer υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 175 και ΙΜΚΟ 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 176 και 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η επόμενη καταπίπτει 179 της κυρίας Γκροστέτ και Ήτρε 5 υπέρ Πρέπει να έλεγξω κάτι πριν. Έχω το 5 και το 6 μαζί. Το ήτρα 6 είναι πιο κάτω. Όχι, το 5 είναι εδώ. ΙΤΡΕ 5 και όχι ητρε 6. 179 λοιπόν και ΙΤΡΕ 5 ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 180 Ζίμπερ με προφορική τροπολογία του εισηγητή και είναι ταυτόσιμο με το ΙΜΚΟ 19. Ναι. Έχετε το προφο... την προφορική τροπολογία στο φακελό σας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το ΙΤΡΕ 5 έχει εγκριθεί. Ναι. Λυπούμε. Δεν έχει νόημα να ψηφίσουμε αυτό το τελευταίο. Καταπίπτουν το 108 και το 90. Πάμε στην 181 και στην 182. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρεις ταυτόσημες. 1.83, 6 ήτρε, 23 employment. Υπέρ. Α, καταπίπτουν, συγγνώμη, κάνω λάθος. Μερικές φορές πέβδω. Και οι επόμενες καταπίπτουν. Τελευταία αιτιολογική σκέψη 46α και β. Τροπολογία Bowies 1.88. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 employment υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 24 κατά. Εγκρίνεται. 26 employment υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. διαδικαστικό της κυρίας Ρον Πέρεντ από την πλευρά της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που παίρνω το λόγο. Θα ήθελα να κάνω μια διακοπή πέντε λεπτών παρακαλώ αν δεν σας πειράζει. Ως πρόεδρος συμφωνώ. Ήταν εξαιρετικά δύσκολη η ψήφιση των τροπολογιών. Να είστε τυπικοί όμως παρακαλώ, να επιστρέψετε σε πέντε λεπτά και όχι περισσότερα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, προχωρούμε. Η κυρία Ντάκμαρ Ροτ Μπέρεντ έχει ζητήσει το λόγο, διότι θέλει να κάνει μια δήλωση. Αλλά θα σας δώσω λίγο χρόνο μέχρι να καθίσετε, για να μπορέσουμε να ακούσουμε προσεκτικά. Παρακαλώ καθίστε. Ντάκμαρ, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι είναι ασυνήθιση η διαδικασία αυτή, ειδικότερα σήμερα που είναι η τελευταία φορά που συνεδριάζουμε. Λυπούμε, αλλά η πολιτική μου ομάδα θα πρέπει να απέχει από την τελική ψηφοφορία. Θέλαμε να μην απέχουμε, αλλά η προσθήκη της νομικής βάσης, το 152 και το θέμα του άρθρου 8.3 είναι πράγματα που σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε. Κάποιες άλλες τροπολογίες μας απορρίφθηκαν, έστω να το δεχθούμε, αλλά αυτά τα δύο δεν μπορώ να τα δικαιολογήσω. Ε, πολύ λυπούμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να απέχουμε από την ε, ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ σαφής η δήλωσή σας. Τώρα λοιπόν θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικό το σχέδιο της πρότασης, όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Ψήφισαν όλοι. Δεν ψήφισαν όλοι. Ψήφισαν όλοι λοιπόν. Πέρα της ψηφοφορίας. 31 υπέρ. 31 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά. 19 αποχές. Ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 31 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, 20 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια σε όλους όσους ε, συμμετείχαν, συγχαρητήρια στους κοιόδης εισηγητές και στο ε, βοηθητικό διοικητικό προσωπικό. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά. Please don't leave. Παρακαλώ μη φεύγετε από την αίθουσα, διότι έχουμε και άλλη δουλειά. Έχουμε να πάμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Σχέδιο συστάσεων του Συμβουλίου για την ασφάλεια των ασθενών. Ε, συμπεριλαμβανομένων και των λοιμόξεων, των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Η συγκήτρια είναι η κυρία Σαρτόρη. Μπορούμε να ψηφίσουμε κατευθείαν ή θέλετε να μιλήσετε. Α, πολύ ωραία. Μπορούμε να ψηφίσουμε κατευθείαν. Εδώ λοιπόν έχουμε τον κατάλογο των, των τροπολογιών και ξεκινούμε την ψηφοφορία των τροπολογιών. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Έχετε όλοι τον κατάλογο ψηφοφοριών μπροστά σας. Παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Τροπολογία υπαριθμών 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές να ψηφίσουμε με το ηλεκτρονικό σύστημα. 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 9 υπέρ 34 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει. 33. Προφορική τροπολογία ΕΛΚ και Σοσιαλιστών. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η εννέα καταπίπτει. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει. 35 της κυρίας Αρτόρη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της τροπολογίας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται επίσης. 38. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Την 37. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. 39 του Μπόουις. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 κατά τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά, άποχες, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 με την προφορική τροπολογία των φιλελευθέρων. Την έχετε ήδη στο φάκελό σας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές. Την 50 ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 της κυρίας Ντάλ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 52 με την τροπολογή την προφολυρική του ΕΛ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 57 υπέρ, 56, να ελέγξουμε την 56, καλώς. Μπορεί να έχω κάνει λάθος. 56 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ποιος είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 10 υπέρ, 32 κατά. Σας ευχαριστώ κυρία Μακίνα. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1 στην αιτιολογική σκέψη 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το σχέδιο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Το ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 50 υπέρ. Κανείς κατά, καμία αποχή. Σχέδιο κανονισμού. Νομοθετικού κανονισμού. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 50 υπέρ, κανείς κατά καμία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, την κυρία Σαρτόρη. Θερμά συγχαρητήρια και σε όλους τους συμμετέχοντες. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλους. Επομένως, προχωρούμε. Πάμε στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Ανάκτηση ετμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού επιβατικών οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων. Οι τροπολογίες εκτείνονται σε τρεις σελίδες. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Αδάμου, ο οποίος αντικαθιστά τον εισηγητή κύριο Παπαδημούλη, αν θέλει να κάνει κάποια δήλωση ή αν μπορούμε να ψηφίσουμε κατευθείαν. Κυρία Αδάμου, έχετε το λόγο. Έχετε εγγραφεί ως αντικαταστάτης του εισηγητή. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Ε, δεν έχω τίποτα να δηλώσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ε, προχωρήσουμε στην ε, ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αρχίζουμε από την τροπολογία υπαρθμών 1. Είσαστε έτοιμοι, έχετε τον κατάλογο των ε, ψηφοφοριών. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε η τροπολογία 1. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 20 υπέρ, κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 20 ήταν υπέρ, 29 κατά. Επομένως απορρίφθηκε. 21 του κυρίου Κρούπα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 22. Ας υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 23. Χάση. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίφθηκε 11 του εισηγητή υπέρ κατά Ας το επαληθεύσουμε. Τροπολογία παριθμών 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. 25 ήταν υπέρ, 22 κατά, εγκρίθηκε. 24 τροπολογία του κυρίου Γιόργενσεν με προφορική τροπολογία εκ μέρους της Γουαϊπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 25 Κόρμπεϊ προφορική τροπολογία της Γκουε κατά Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. 28 ήταν υπέρ, 19 κατά. Ε, είχε εγκριθεί. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 26 του Μάρτιν Κάλαναν με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Λίγες 20 τα χέρια του. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. 41 υπέρ, 5 κατά και μόνον δύο αποχές. Σαφέστατα ήταν υπέρ. Λοιπόν, δεκαετία του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίφθηκε. 27 υπέρ, κατά, αποχές. Ας το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. 27 μπούζεκ του Γέρτζι Μπούζικ. Πέρα της ψηφοφορίας, 32 υπέρ, 18 κατά, 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε, 29 υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, επαληθεύουμε την 29. Ζήμπερ. Πέρασε τη ψηφοφορίας. 21 ήταν υπέρ, 28 κατά. Απορρίφθηκε. 30. Του ιδίου εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 14. Θα ψηφίσουμε δύο τμήματα ξεχωριστά. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τώρα το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 15. Θα ήθελα να ελέγξω το δεύτερο τμήμα της 14. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας. 15 ήταν υπέρ και 35 κατά. Είχε Λοιπόν, τώρα 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 18 έχουμε μια προφορική τροπολογία της ολιστικής ομάδας υπέρ κατά Αποχές εγκρίθηκε. Λοιπόν, τροπολογία 2 του εισηγητή υπέρ κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 3 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 4 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Η 5 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 6 με μία προφορική τροπολογία της ΓΚΟΥ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Ας το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Επαληθεύουμε την 7 του εισηγητή. Πέρασες τροπολογία. ψηφοφορία. Ήταν 28 υπέρ 22 κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 9 υπέρ κατά. Θα το ελέγξουμε η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας 27 ήταν υπέρ, 23 κατά. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και τώρα θα βάλουμε το σχέδιο της έκθεσης σε ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 46 ήταν υπέρ. Ένας κατά, τρεις αποχές. Ο Ανδρέας έκανε μια πολύ καλή πρόταση. Ε, πριν να φύγουμε και να εξαφανιστούμε, ε, να φωτογραφηθούμε. Μας περιμένει έξω ο φωτογράφος ε, Λοιπόν, εντάξει, αλλά θα πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε το σχέδιο της έκθεσης, όπως είπαμε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, 42 ήταν ε, υπέρ, ε, ένας κατά, τέσσερις αποχές. Συγχαρτήρια στον κύριο Παπαδημούλη, τον εισηγητή. Ελπίζω ότι ο κύριος Αδάμου θα διαβιβάσει και θα ενημερώσει τον εισηγητή για το εξαίρετο αυτό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Και τώρα αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, ας βγούμε όλοι μαζί και ας βγάλουμε μια φωτογραφία. Λοιπόν, μας περιμένει έξω από την αίθουσα ο φωτογράφος, επομένως πρέπει να μεταφερθούμε έξω. Παρακαλώ.